Αγαπητοί, αγαπητοί συνάδελφοι, άρχεται η συνεδρίαση εκ νέου. Τα πρακτικά της χτεσινής συνεδρίασης ήδη σας έχουν διανεμηθεί. Δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει. Δεν βλέπω να θέλει κάποιο να υποβάλει παρατηρήσει. Κατά συνέπεια θα εγκριθούν τα πρακτικά. Ακολουθούμε στη συνέχεια την ημερήσια διάταξη με δήλωση της Επιτροπής για τον σεισμό στην περιοχή των